Ε, Καλημέρα σε όλους σας. Ακόμα δεν έχουμε ε, απαρτία. Δεν ξέρω, θέλετε να περιμένουμε λίγο. Γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα να καλύψουμε. Θα σας πρότεινα να αρχίσουμε. Διότι... μέχρι τις 9.30 πρέπει να έχουμε τελειώσει ε, τα πρώτα θέματα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το διευρυμένο προεδρείο που προβλέπεται να συνεδριάσει στις 11 και 4 ακυρώθηκε. Γιατί απουσιάζουν πάρα πολλοί συντονιστές. θα συσταθεί η Διευθυντική Επιτροπή για να δούμε ποια θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου για τις κατεξουσιοδότηση πράξης ε, για τις σχέσεις μας για την Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Οι εκπρόσωποι ε, της Επιτροπής μας ε, αυτό προσκαλούνται να συμμετέχουμε. Από το 2005 κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις και ζήτησα από τον κύριο Μπροκ να με εκπροσωπήσει εκεί και την Επιτροπή μας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσει του Πρόεδρου που θα σας κάνω και έρχομαι στο επόμενο θέμα που είναι συμφωνία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Και το σημείο 4 ταυτόχρονα σε σχέση με την επανεισδοχή ε, παρανόμως διαμενόντων, επαναπρόθεση καλύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω ε, το λόγο στον κύριο Λίζεκ. Ευχαριστώ. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και εδώ και στην Ολομέλεια. Εχθές, πολλοί συνάδελφοι και από τη δική μας επιτροπή είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κύριο Σακασφίλη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες αυτό τον καιρό. Και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μερικά ζητήματα. Ο Γεωργιανός ε, Πρόεδρος εξήρε την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτές τις δύο συμφωνίες. Στην Επιτροπή Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, που είναι αρμόδια επί της ουσίας συζητούν αυτό το θέμα της επαναπροώθησης ε, προσώπων που διαμένουν στις χώρες μας παράνομα, καθώς επίσης και ένα σύστημα διευκόλυνσης θεωρήσεων ε, διαβατήριων. Τέλειο Οκτωβρίου μάλλον θα έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση για τις βίζες. Στις 23 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, άκουσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Ελευθεριών θα εγκρίνει το κείμενο στις 25-26 Οκτωβρίου. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία το Δεκέμβρη στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε για τις δύο αυτές εκθέσεις. Ε, επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικές πληροφορίες τώρα. Στις 17 Ιουνίου Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία υπέγραψαν συμφωνία για διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου. Το θέμα είναι να μειωθούν τα τέλη και να διευκολυνθούν ε, οι γεωργιανοί πολίτες στις μετακινήσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. από 60 ευρώ που έκανε η Visa τώρα θα κάνει 35 και ε, δικαιούνται Visa και άλλες κατηγορίες γεωργιανών πολιτών. Τον Οκτώβριο του 2010 θα υπογραφεί συμφωνία και το 2011 θα τεθούν σε ισχύ και οι δύο συμφωνίες αφού ε, κυρωθούν από τη Βουλή της Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2008 άρχισαν διαπραγματεύσεις για τη θεωρήση διαβατήριων. Για την απελευθέρωση δηλαδή και την διευκόλυνση που μας απασχολεί τώρα. Και βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστούν στα πλαίσια της πολιτικής της γειτονίας, όπως λέγεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επαναπροώθηση των προσώπων που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να ενισχύσουμε ε, τη συνεργασία μας με τη Γεωργία να καταπολεμήσουμε την λαθρομετανάστευση. Θέλουμε να επιταχυθούν οι διαδικασίες για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων ε, που ελέγχονται και ε, να διαπιστώνονται πιο εύκολα οι παράτυποι μετανάστες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο, διότι το πρόβλημα της επανεισδοχής με τη Γεωργία δεν είναι μεγάλο μεν, η Γεωργία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια χώρα που έχει συμφωνίες και υπογράφει συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και έχει υπογράψει και ε, τη συμφωνία για το καθεστώς του πρόσφυγα. Και είναι και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης η Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την ευκόλυνση θεώρηση διαβατηρίων και αυτή νομίζω ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ γρήγορα και θα τεθεί γιατί έτσι έχουμε καλύτερες επαφές και πολιτιστικές και οικονομικές και ανθρώπινες και συσφίγουμε τις σχέσεις μας και τους δεσμούς μας με τη Γεωργία. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το 2007 υπογράψαμε μια συμφωνία οι πολίτες της Απχαζίας και της Νότιας Ουσιατίας που έχουν ε, ρωσικά διαβατήρια. είναι σε ε, καλύτερη, ευνοϊκότερη θέση από τους υπόλοιπους, από τους πολίτες που δεν έχουν ρωσικό διαβατήριο. Και ελπίζω αυτή η συμφωνία να ε, υπογραφεί σύντομα και να βελτιωθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή και στις σχέσεις μας με τη Γεωργία. Και οι διαπραγματεύσει νομίζω βαίνουν καλώ. Λοιπόν, με βάση όλα αυτά που σα είπα, παρακαλώ να εγκρίνετε τη γνωμοδότησή μου και σα ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο να πάρει το λόγο, όχι. Κανένα από του συναδέλφου ε, δεν θέλει να παρέμβει. Οπότε, ίσω μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αν είναι στην αίθουσα. C'è un consulto in atto, lo dico per i colleghi che non stanno vedendo tra i dirigenti della Commissione, Λοιπόν, δεν φαίνεται να είναι εδώ ούτε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ε, α, όχι, κάποιο είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπερνάρ Φιλίπ ονομάζομαι. Να σα πω σύντομα δύο-τρία πράγματα. Αυτό το θέμα της διευκόλυνσης θεώρησης και επανεισδοχής αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Υποστηρίζουμε αυτή τη βασική ιδέα προσέγγισης των πληθυσμών. Γνωρίζουμε βεβαίως επίσης την ανάγκη που υπάρχει γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να βοηθηθεί η Γεωργία μετά τον πόλεμο να ανοικοδομηθεί και να αναδομηθεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό λοιπόν και όπως ήδη υπόθηκε στην προηγούμενη παρέμβαση ε, γνωρίζουμε, είμαστε μάλλον ε, ε, πεπισμένη για την κατάσταση της δημοκρατίας και των ε, συνθήκων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γεωργία. Έχει υπογράψει η Γεωργία διάφορες συμβάσεις μεταξύ των οποίων αυτή για τους πρόσφυγες του 1951 και να σας πω ότι έχουμε μια, ένα συνεχιζόμενο διάλογο στα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Γεωργία που είναι εξαιρετικά θετικός. Μάλιστα είχαμε τρεις συνόδους διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Γεωργία και άρα... Ε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ποιότητα του διαλόγου και στη δυνατότητα ε, εάν υπάρξουν προβλήματα να αναφερθούν αυτά τα προβλήματα σε ελεύθερο και ανοιχτό πλαίσιο με την γεωργιανή πλευρά. Είμαστε λοιπόν πολύ υπέρ των προόδων που έχουν σημειωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλετε κάτι ακόμα να πείτε? Θέλετε να μας πείτε πώς λέγεστε? Ναι, ευχαριστώ. Ντίτριχ Πάλμερ. DG Home. Αυτέ οι δύο συμφωνίε θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν μπορεί να αρχίσει να ισχύει η συμφωνία περί θεωρήσεων πριν από την συμφωνία περί επανεισδοχής. Νομίζω πως αυτό κατέστη απόλυτα σαφές κατά την παρουσίαση του εισηγητή. για την επανεισδοχή είχαμε, ε, είχαμε ένα προβληματάκι γιατί αυτή η ε, συμφωνία δεν είχε συνυπογραφεί ακόμα. Είναι κάπω πρόημο λοιπόν να το συζητάμε γιατί δεν είχε ακόμα υπογραφεί λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και την Ιρλανδία και τις σχετικές θέσεις τους. Ε, αλλά απειλείονται αυτά κατά τη διάρκεια της σημερινή μας ε, συνομιλίας και ελπίζουμε πως σύντομα θα υπογραφεί η συμφωνία αυτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τότε θα μπορέσουμε να υπογράψουμε και εμείς και να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτήν την περαιτέρω διευκρίνηση. Εγώ θα δώσω το λόγο για τα τελικά σχόλια στον εισηγητή μας, τον κύριο Λίζε, που είναι φυσικά... Εκείνος που θα συνοψίσει. Όχι, δεν θέλετε. Ωραία. Dario ε, μάλιστα, αυτό έχουμε το χρονοδιάγραμμα για την πρώτη εξέταση του σχεδίου που ήδη έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου. Σήμερα δηλαδή. Έχουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 20 του μηνός και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα ε, γίνει στις 5 Οκτωβρίου. A questo punto, siccome i relatori non vedo, eh, siamo stati <laughs> Eh, λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή για πέντε λεπτά περιμένοντας ε, την άφηξη των εισηγητών για την δημόσια κρόση για την ευρωπαϊκή στρατηγική στην Μαύρη Θάλασσα. Σε 5 λεπτά τα ξαναλέμε.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

Περιμέναμε λίγα λεπτά για να έχουμε κάποια... την απαραίτητη εκπροσώπηση των συναδέλφων. Δεν έχουμε ακόμα απαρτία, αλλά πιστεύω πως οι προσκεκλημένοι μας είναι όλοι εδώ και οι εισηγητές μας, οι οποίοι ήταν στην ώρα τους να καλωσορίσω τους εισηγητές, τους προσκεκλημένους μας, τους ομιλητές μας, τους εισηγητές μας και όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Στατικική για τη Μαύρη Θάλασσα είναι μια στατικική που σκοπό έχει να ξεκινήσει μια συζήτηση για την περιφερειακή συνεργασία στην Μαύρη Θάλασσα και στον ε, ρόλο μας ε, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και γι' αυτό και θεωρήσαμε πως ήταν σκόπιμο να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει για τις εκθέσεις, την έκθεση του συναδέλφου Ρεάνου για αυτό το θέμα. Έχουμε τον δόκτορα Μίν Κέφε που είναι εξέχουσα προσωπικότητα του, του Ινστιτούτου για τις Διεθνείς ε, και ε, Σπουδές της Σόφιας, την κυρία Δελκούρ που είναι από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικής του Παρισιού και τον δόκτορα Μάρκα Κάνιχαμ του Black Sea Trust του German Marshall Fund να καλωσορίσω και τους εισηγητές που είναι υπεύθυνοι για γνωμοδότηση, διεθνείς υποθέσεις, βιομηχανία και έρευνα και περιφερειακή πολιτική, ε, ε, επιτροπές που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για να συμβάλλουν στη συζήτηση με γνωμοδοτήσεις. Να δώσω αμέσω το λόγο στον συνάδελφο για να παρουσιάσει το θέμα. Το συνάδελφο Ουγγουρεάνου. Σας ευχαριστώ όλους. Καλωσορίζω τους διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας, κύριο Αλμπερτίνη, σήμερα, καθώς και τη γραμματεία της ΑΦΕΤ για την διοργάνωση της παρούσας ακρόασης, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός νέου οράματος σχετικά με την περιοχή της ε, Μαύρης Θάλασσας και που θα μας δώσει τη βάση, θα μου δώσει τη βάση για τη σύνταξη της εκθέσεώς μου. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους με ικανοποιεί η σημερινή ανταλλαγή απόψεων και ο πρώτος λόγος, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει καλή αφετηρία για τις συζητήσεις μας, είναι η στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και για τις προμήθειες ενέργειας. Από το 2007, με την ένταξη της Ρουμανίας και Βουλγαρίας, η Μαύρη Θάλασσα έγινε εν μέρη, εσωτερική θάλασσα της Ένωσης. Τα όσα συμβαίνουν λοιπόν επί της Μαύρης Θάλασσας και γύρω από αυτήν, έχει τώρα πια άμεση συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο αυτό εισήγαγε και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Μαύρη Θάλασσα. Πώς αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσέγγιση αυτή ε, με το σύνολο των θεμάτων της Μαύρης Θάλασσας. Η καλύτερη πολιτική θα ήταν να επιτρέψουμε στη Μαύρη Θάλασσα να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο. Θα συμφωνήσετε. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι η Ένωση ανεγνώρισε την στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας το 2007 ξεκινώντας την πρωτοβουλία της συνέργειας της Μαύρης Θάλασσας. Και η ιστορία της, η έλλειψη ιστορίας της είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η σημερινή ακρόαση. Η Black Sea Synergy υποτίθεται ότι θα δημιουργήσει ένα χώρο σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας. Ακεί όμως αυτό. Και τι επέτυχε μέχρι τώρα η συνέργεια αυτή, η συνεργασία αυτή για τη Μαύρη Θάλασσα. Εμείς νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι, θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής διότι έφτιαξε μια συγκεκριμένη αντίληψη γύρω από την Μαύρη Θάλασσα και για τη σημασία της, τα δική της σημασία. Αλλά τώρα τρία χρόνια μετά από την σύλληψη αυτής της ε, ιδέας τα αποτελέσματα είναι ακόμα αμφισβητούμενα. Το 2008 η Κομισιόν εξέδωσε έκθεση για την, την πρώτη χρονιά εφαρμογής της Black Sea Synergy. Αλλά το 2009 και 2010 πέρασαν τα δύο αυτά χρόνια και δεν προέκυψε άλλη έκθεση τέτοιου είδους. Όπως κάποιος μου λέει εδώ και πολύ ε, σοφά, ίσως να μην υπήρξαν άλλα επιτεύγματα. Να το συζητήσουμε. Στο μεταξύ όμως, οι προκλήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας εξακολουθούν να υπάρχουν. Και μάλιστα ορισμένες από αυτές εξελίχθηκαν και έφτασαν να γίνουν σημαντικές κρίσεις. Ο πόλεμος Γεωργίας-Ρωσίας τον Αύγουστο 2008. Βάθινε τις προκλήσεις αυτές. Η η ιστορία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και η παρουσία του που θέτει, ε, προκαλεί σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια. Η ενεργειακή κρίση με συμμετοχή της Ρωσίας συνεχίζεται. Ορισμένες από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας παρουσιάζουν ανησυχητικές τάσεις κάποιων αυταρχικών πολιτικών. Υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα ορατότητας δηλαδή για το Black Sea Synergy. Και προσθέτω ευθύ αμέσω ότι δεν έγιναν υπουργικέ διασκέψεις υψηλού επίπεδου πρόσφατα. Ένα άλλο πρόβλημα που βλέπω είναι η ξεκάθαρη δημοσιονομική πρικοδότηση της πολιτικής της ε, συνέργεια τη Μαύρη Θάλασσας. Συνοψίζοντας, θα πω ότι υπάρχει σήμερα αδύρυτη ανάγκη να αναβαθμιστεί η συνέργεια Μαύρη θάλασσα και να ενταχθεί στη στρατηγική της Ένωσης, βασιζόμενη στην εμπειρία που διαθέτουμε της πρόσφατης Ανάπτυξη της στρατηγικής της Ένωση για τη Βαλτική θάλασσα. Έχουμε λοιπόν τώρα τη Synergy, αλλά δεν έχουμε τη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή ποια πλονεκτήματα θα προσφέρει, ποια ωφελήματα θα αποφέρει. Μια πλήρη στρατηγική θα σήμαινε μια συνολική προσέγγιση της Ένωσης για την περιοχή αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με ξεκάθαρους στόχους, με πρωτοβουλίες και με benchmarks, με κριτήρια δηλαδή επιτυχίας. Επίσης, μια ειδική γραμμή στον προπολογισμό, ένα ειδικό κονδύλι δηλαδή, για τη στρατηγική αυτή. Με λίγα λόγια, εκεί βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ανυπομονώ να ακούσω τις τοποθετήσεις των εμπειρογνωμών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκουρεάνο, το λόγο έχει ο πρώτος προσκεκλημένης μας, ο, ο δόκτωρας Όνιαν Μίνκεφ από το Ινστιτούτο Περιφερειακών και Διεθνών Σπουδών της Σόφιας. 10 με 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ε, Πρόεδρε, ε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, η περιοχή της ε, μαύρης θάλασσας μας ανησυχεί όλο και περισσότερο για λόγους ασφαλείας και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, στρατηγική αναδιάθρωση στην περιοχή είναι η δεύτερη τα τελευταία 20 χρόνια μετά τη μετάβαση από τον κομμουνισμό και τη μετασοβιετική ε, περίοδο που οι περισσότερες ανατολικές χώρες στράφηκαν στις ευρωατλαντικές δομές ασφάλειας ε, από πλευρά αξίας θεσμών και χεγγύων για την ασφάλειά τους, τώρα έχουμε σε κάποιο βαθμό την αντίστροφη διαδικασία. Η Ρωσική Ομοσπονδία και οι παραδοσιακοί παράγοντες της περιοχής, η Ρωσία λοιπόν και η Τουρκία, προσπαθούν να ανακτήσουν μερική επιρροή σε κάποιες χώρες της περιοχής. Και αυτή η αναδιάρθρωση είναι βασική ανησυχία ασφάλειας, γιατί οποιαδήποτε στρατηγική αναδιάρθρωση θέτει τρία βασικά ζητήματα ασφαλείας. Το πρώτο είναι το ζήτημα των συνόρων, των στρατηγικών ισορροπίων, δηλαδή το δεύτερο είναι των κοινοτήτων και των σχέσεων μεταξύ τους και κοινοτικά ίσως προβλήματα και συγκρούσεις ίσως προς το status quo των κοινοτήτων και το τρίτο είναι η θεσμική αδυναμία γιατί η στρατηγική αναδιάρθρωση σημαίνει και αναδιάρθρωση των ελίτ, των θεσμών και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Υπάρχουν ε, διάφορα πρότυπα ασφάλειας. Το πρώτο είναι το ευρωατλαντικό πρότυπο, το ευρωπαϊκό μοντέλο αλληλεξάρτησης και δημοκρατίας στις διεθνείς σχέσεις και στις ε, διευθετήσεις για την ασφάλεια. Δυστυχώς το μοντέλο αυτό, το πρότυπο αυτό, τα τελευταία 5-7 ε, χρόνια υποχωρεί. Το δεύτερο πρότυπο είναι αυτό που επιβάλλουν status quo μεγάλες δυνάμεις του 19ου αιώνα και αυτό σήμερα εκπροσωπείται ε, από τη σημερινή Ρωσία και όλο και περισσότερο από τη σημερινή Τουρκία. Και μετά υπάρχει το πρότυπο των νεοσύστατων κρατών ε, στις περιοχές εκεί που ε, είναι σε μια διαδικασία οικοδόμησης κράτους και θέλουν να θέσουν τη νέα τους ανεξαρτησία μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωατλαντικά δεδομένα. Και κάτι άλλο που δεν είναι ίσονο σημασία και δυστυχώ νέο παράγων που αυξάνεται και θα αποκτήσει έτσι πολύ μεγάλη σημασία στην εξίσωση ασφαλεία τη περιοχή εκεί, που είναι ο ακραίο Ισλαμικό αποσχιστικός παράγων ε, που παρατηρείται όλο και περισσότερο. Έχουμε λοιπόν στρατηγική μετατόπιση από μία ισορροπία δυνάμεων σε μία άλλη ισορροπία δυνάμεων. Και έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε διάφορα βασικά στοιχεία ασφαλείας στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Πρώτον, η στρατιωτική ασφάλεια. Λίγα είναι τα θετικά που θα μπορούσαμε να πούμε εκεί. Δυστυχώς, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη στρατικοποίηση της περιοχής. Έχουμε ε, νέες βάσεις της Ρωσίας στην Απχασία και στη βόρειο αιτία της αποσχιστής περιοχές και νέες τουρκικές βάσεις, μία βάση προκειμένου στη δυτική επαρχία του Αζερβαϊτζάν στα σύνορα με την Αρμενία στο νότιο Κάφκασο αμυντική κούρσα σε όλες τις χώρες αλλά ιδιαίτερα στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία αυξάνεται η ισόρευση όπλων, οι εξοπλισμοί, ε, ε, στρατιωτική δύναμη, οι ένοπλες δυνάμεις και οι λεγόμενες παγωμένες σειράξει μέχρι τώρα έχουν αθερμαθεί. δηλαδή Απχασία, ε, Νότια Οσετία και Ορεινό Καραμπάχ. Αυτή η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη, γιατί μπορεί να οδηγεί σε πλήρη απόψυξη εντό αγωγικών, αθέρμαση των συγκρούσεων στην περιοχή και μπορεί να εμφανιστούν και ένοπλες σειράξει που βεβαίως επηρεάζουν και τις θέσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Στη συνέχεια, το είπα και προηγουμένω. επαναλαμβάνονται οι σειράξει μεταξύ εθνοτήτων και κοινοτήτων, όχι μόνο στο Νότιο Κάφκασο, αλλά ξανανοίγουν τα προβλήματα με την υπερνηστερία και τη Μολδαβία εμφανίζονται πολύ έντονες και ατυχείς διαδικασίες αποσχιστικών τάσεων ακραίων στο Βόρειο Κάφκασο και αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από κανέναν ούτε η Ρωσία ούτε άλλες χώρες της περιοχής, ούτε οι δυτικοί σύμμαχοι δεν θα μπορούσαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα μέχρι τώρα για να καταφέρουν να πλαισιώσουν, να περιορίσουν αυτές τις τάσεις που εμφανίζονται και τις αποσχιστικές πιέσεις και να τις έσουν εντός ενό πλαισίου ε, που θα δίνει ένα ορίζοντα για πιο ασφαλή ε, περιοχή στο μέλλον. Επόμενο στοιχείο, η ε, ναυτιλιακή ασφάλεια. Ουσιαστικά οι χώρες του status quo εκεί, η ε, Ρωσία και η Τουρκία έχουν ε, ναυτική ε, συνηγεμονία στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό είναι σημαντικό και για την Τουρκία αλλά και για τη Ρωσία που ανανέωσε τη συμφωνία της με την Ουκρανία για την παρουσία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Και όπως γνωρίζουμε σύμφωνα με τη σύμβαση του Μόντρεαλ δεν μπορούν άλλες δυνάμεις να μπουν στον εύξον πόντο για περισσότερο από τρεις εβδομάδες ναυτικό άλλης χώρας δηλαδή και θα Έπρεπε να ρωτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποψήφια χώρα Τουρκία όταν και αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία και θα ισχύει και η ΚΕΠΑ κατά κάποιο τρόπο θα συνιστά εξαίρεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πολεμικό ναυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα γίνει με τη σύμβαση του Μόντρεαλ γιατί εξ όσων γνωρίζω αυτό είναι και ένα τμήμα της ΚΕΠΑ. Η ναυτική ασφάλεια ε, στη Μαύρη Θάλασσα συνδέεται στενά με την ναυτιλιακή ασφάλεια και έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ε, με την αυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα ακόμα και αν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο βελτίωσης ε, των ε, επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη Μαύρη Θάλασσα, στην πράξη αυτό δεν το βλέπουμε. Τα τελευταία χρόνια τρία πλοία βυθίστηκαν δύο-τρία μίλια από τις ακτές της Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ουκρανίας χωρίς καμία σοβαρή απόπειρα από πλευράς των αρχών των κρατών αυτών ε, έρευνας και διάσωσης ε, του πληρώματος ή του πλοίου με μικρές εξαιρέσεις. Οι περισσότεροι ναύτες ε, πνίγηκαν. Υπάρχει επίσης κάτι πολύ σημαντικό υπάρχουν ζητήματα εκεί ναυτιλιακής ασφάλειας ε, που συνδέονται περισσότερο και με τους ελέγχους των συνόρων για το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, δουλεμπόριο κτλ. και λαθρεμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θετική πείρα από την αποστολή ε, στη Μολδαβία και την Ουκρανία για τη βοήθεια στον έλεγχο των συνόρων και επίσης ε, ε, έχει τα τελευταία χρόνια συλλέξει εμπειρία από την παρατήρηση στη Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσει τις δυνάμεις της και να τις εντείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει βέβαια μέσα σε ένα θετικό πολιτικό πλαίσιο της χώρας της περιοχής έτσι ώστε τα σύνορα φυλάσσονται με το σωστό τρόπο και ιδιαίτερα στο Βόρειο Κάυκασο να μην επιτρέπει να εμφανίζονται μαύρες κοιλίδες όπου ευνοείται το λαθρεμπόριο ναρκωτικών προς δυσμάς και πυρηνικής τεχνολογίας προς Ανατολάς κτλ. Η ενεργειακή ασφάλεια τώρα ένα θέμα πάρα πολύ δημοφιλές και εγώ ίδιο δεν θέλω να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε για την ενεργειακή ασφάλεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα εφοδιασμού και ασφάλειας τη ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης, συνδέονται με τη στρατηγική τη Ρωσική Ομοσπονδία, που προσπαθεί όσο περισσότερο, αν μπορεί, να έχει καθεστώ μονοπωλιακό ε, να είναι ο μοναδικός προμηθευτής ενέργειας δηλαδή στις χώρες κεντρικής και ανατολικής ε, περιφέρειας της Ευρώπης. Αυτό έχει και πολιτικές συνέπειες και βεβαίως οικονομικές και επιχειρηματικές διότι το μονοπόλιο σημαίνει ακριβές τιμές ε, υψηλές τιμές και έχει και επιπτώσεις στην ασφάλεια. Όχι μόνο από πλευράς αφηρημένης, κάποια μελλοντική στρατηγική κατάσταση, αλλά και με βάση τα σημερινά δεδομένα ότι αυτό το είδος στο μονοπόλιο ασκείται μέσω εντατικών επαφών μεταξύ των ολιγαρχών στη Ρωσική ε, Ομοσπονδία που ελέγχουν την ενέργεια και ε, τα γειτονικά κράτη και στο μετασοβιετικό χώρο ας πούμε. Οπότε μέσω αυτής της στρατηγικής που θέλει η Ρωσία να μονοπολεί την αγορά ενέργειας, βλέπουμε ότι ε, αυξάνονται οι φαιές ζώνες στην οικονομία, στην Ανατολική Περιφέρεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και από την οπτική που σήμερα έχει καθορίσει για τον εαυτό της Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μαύρη Θάλασσα, μπορούμε να τονίσουμε πρώτον τη διασυνοριακή συνεργασία έτσι ώστε να βελτιωθεί ε, αυτή η θεσμική συνεργασία με τις χώρες του ευξήνου πόντου που όπως σας είπα αφορά την Ευρώπη, στο λαθρεμπόριο, στη μετανάστευση, στις φαίες Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, συμμετέχει περισσότερο σε ναυτιλιακές και ναυτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, έρευνα και διάσωσης. Και ένα τελευταίο που είναι και σημαντικό όμως, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιβαλλοντική ασφάλεια. Στο Βόσφορο, ας πούμε, έχουμε προβλήματα, θα περάσουν νέοι πετρελαγωγοί από εκεί που μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Η πολιτική λοιπόν ραχοκοκαλιά αυτών των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ήταν να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία όχι μόνο προσέγγιση τώρα προσμά όπως λέγεται διεθνώς αλλά και με άλλους τρόπους με σταθεροποίηση των σχέσεων που να βασίζονται σε αρχές και αξίες έτσι ώστε να έχουν και μια πιο μακροπρόθεσμη πρόπτικη Και επίσης να ε, προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει τις πολιτικές του δεύτερου σημαντικού πρωταγωνιστή και της Τουρκίας που είναι και υποψήφια προς ένταξη χώρα και που τελευταία ε, λίγο απομακρύνεται από τις ευρωατλαντικές δομές και ασφάλειες και από πλευράς αξιών και αρχών αλλά και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, δόκτωρα Μίνκεφ. Το λόγο έχει η δόκτωρα Λόρντελ Κούρα. Σας ευχαριστώ. Η δική μου εισήγηση θα εστιάσει στην ε, συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας και πιο συγκεκριμένα σε τέσσερα κύρια σημεία. Καταρχήν λοιπόν θα αναφέρω εν συντομία τους παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία της ε, συνεργασίας της για την Μαύρη Θάλασσα. Θα σας δώσω μια γενική εικόνα της εφαρμογής αυτής της ε, συνεργασίας το μικρόφωνο της ομιλήτριας δεν λειτουργεί δυστυχώς. By Πώς λοιπόν ε, επηρεάζεται από το τοπικό πλαίσιο η διεθνής αυτή συνεργασία και τέλος θα προτείνω κάποιους τρόπους για βελτίωση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής συνεργασίας τρεις παράγοντες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην κίνηση της ε, συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Καταρχήν, μεγαλύτερη προσοχή δόθη στην ε, περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ένωσης προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία το 2007 Δεύτερον, αυτό το νέο κύμα διεύρυνση σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευρωπαϊκή ανησυχία για την ασφάλεια ανεφοδιασμού σε ενέργεια οδήγησε σε μεγαλύτερη εμπλοκή σε μια περιοχή που μέχρι στιγμής είχε μείνει στο, στο παρασκήνιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, η συνεργασία αυτή ξεκίνησε και μέσα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής γετνίασης και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ε, χλιαρής αξιολόγησης αυτής της ε, πολιτικής γυπνίασης όσον αφορά θέματα ασφαλείας κυρίως. Σε αυτό το πλαίσιο η περιφερειακή συνεργασία θεωρήθηκε απαραίτητη ώστε να συμπληρώσει την διμερή διάσταση που μέχρι στιγμής είχε επικρατήσει στην πολιτική γυπνίασης. στην πρόταση λοιπόν της Ευρώπης και της Κομισιόν, η, το 2007 ξεκίνησε επισήμως η συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας σε μια συνάντηση που, των Υπουργών Εξωτερικών στο Κιέβο το 2008. Ε, αποφασίστηκε ως ένα ευέλικτο πλαίσιο ή εν πάση περιπτώσει μια γενική πολιτική που συμπληρώνει τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η πολιτική γυτνίασης, η πολιτική Ένταξη απέναντι στην Τουρκία αλλά και η συνεργασία με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, επίσης σχεδιάστηκε ως μια κοινή προσπάθεια, ένα κοινό εγχείρημα όπου θα συμμετείχαν όλοι οι περιφερειακοί ε, φορείς και οργανισμοί η συνεργασία αυτή προβλέπεται για την, προβλέφθηκε μάλλον για την ενίσχυση της σταθερότητας και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Προς αυτό το σκοπό, τα έγγραφα που προτίμασαν οι υπηρεσίες της Κομισιόν περιλάμβαναν διάφορους ε, στόχους προτεραιότητες που πήγαιναν από την παιδεία, στη χρηστή διακυβέρνηση, ε, στην αλληλεία ή το περιβάλλον. Η έκθεση για την συνεργασία και την, πρώτο, πρώτη έκθεση μάλλον για την εφαρμογή της συνεργασίας αυτής ε, έδειξε περιορισμένες, περιορισμένα επιτεύγματα και λιγοστή πρόοδο με σχεδόν καθόλου πρόοδο για τα πολιτικά και θέματα και τα θέματα ασφάλειας. Η δημιουργία τομεακό και συνεργασία σε τρεις ε, τομείς κλειδί, μεταφορές, ενέργεια, και περιβάλλον. Το περιβάλλον, ή μάλλον η συνεργασία για το περιβάλλον ξεκίνησε νωρίτερα φέτος. Και δεύτερον, δεύτερη εξέλιξη ήταν η διασυνοριακή συνεργασία. Ε, έγιναν, ε, έγινε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας και δόθηκαν 17,5 ευρώ το, μέχρι το 2013. Ωστόσο η διαδικασία επιλογής των προγραμμάτων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μια άλλη σημαντική πτυχή στην εφαρμογή της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα είναι η συνεργασία με άλλες χώρες εταίρους στην περιφέρεια αλλά και με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς. Από το 2007 η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, ε, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου όπου γίνονται τακτικές συνεδριάσεις. Ωστόσο, ο διάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή στη συνεργασία με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, υπάρχει πεδίο για συνεργασία με το Φόρουμ της Μαύρης Θάλασσας. Μια τέτοια συνεργασία όμως δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Όλα αυτά συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν εφαρμοστεί. Γενικώ η συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα έχει επηρεαστεί αρνητικά από διεθνείς ε, και περιφερειακές εξελίξεις αλλά και από τις εξελίξεις στην Ένωση. Σε διεθνές επίπεδο μέχρι το 2009 Λόγω των σχέσεων μεταξύ των δύσκολων σχέσεων ΙΠΑ ε, και Ρωσίας, το θέμα της Μαύρης Θάλασσας ε, είχε επηρεαστεί. Τα τελευταία δύο χρόνια η Προεδρία, τα κράτη-μέλη και τη οι θεσμοί της Ένωσης βασικά σχολιόνταν με την επικύρωση της ε, συνθήκης Λισαβόνας και με την οικονομική κρίση. Ε, ταυτόχρονα οι ανατολικές πολιτικές της Ένωσης βασικά ε, καθορίστηκαν από την ανατολική συνεργασία που σε μεγάλο βαθμό επισκίασε τη συνεργασία με τη Μαύρη Θάλασσα. Σε περιφερειακό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε την προσέγγιση της Ρωσίας στην ε, Μαύρη Θάλασσα που τη θεωρεί δικό της ε, μπαϊράκι και ε, στην έλλειψη αποτελεσματικότητας των πολλών φορέων. Και ωστόσο το πλαίσιο είναι ρευστό και έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τώρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την Ένωση και για αυξημένη συνεργασία. Από τη μια πλευρά Η Ουκρανία και η Τουρκία έχουν στραφεί πιο κοντά προς την Ρωσία, ενώ από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μεγάλο εταίρο και για τις δύο αυτές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης φαίνεται να είναι το, το κέντρο βάρους της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες. Τώρα, πιθανή τρόποι για να προχωρήσουμε. Θα... Υπάρχει έλλειψη πολιτικής συνεργασίας, υπάρχει η έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών, ε, μηχανισμών πολιτικών, η έλλειψη ορατών δημοσιονομικών πόρων, η συνεργασία αυτή χρηματοδοτείται από διάφορους πόρους, ε, περιφερειακή πολιτική, MPI και το, μέσο, το προενταξιακό μέσο, έλλειψη επίσης ε, βασικών πρωτοβουλειών με, με ανατολικούς εταίρους και όπως δείχνει και το παράδειγμα της διασυνορικής συνεργασίας, ο αργός ρυθμός στον αντοπισμό την αξιολόγηση και την εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων. Ερώτηση λοιπόν, αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με τη Μαύρη Θάλασσα ακόμα σήμερα. Κοιτάξτε, από τη μια πλευρά υπάρχουν έντονα αιτήματα για περιφερειακή συνεργασία, για παράδειγμα, όταν αφορά τα περιφερειακά δημόσια αγαθά όπως το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά αυτά τα κίνητρα για την περιφερειακή συνεργασία υπονομεύονται από τα θέματα ασφάλειας, όπως ε, περιφερειακές συγκρούσεις για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα κατά πόσο η συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα είναι ακόμα επίκαιρη σήμερα, εμείς απαντούμε πως ναι, γιατί ε, συμπεριλαμβάνει ε, και εμπλέκει όλους τους περιφερειακούς παίκτες συμπεριλαμβανομένες της Ρωσίας και της Τουρκίας. Έτσι, η συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα έχει μεγαλύτερο δυναμικό για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες που διαφορετικά τοποθετούνται σε διαφορετικά πλαίσια πολιτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η συνεργασία αυτή μπορεί να παίξει ένα καλό ρόλο για τη διευκόλυνση των, γειτονικών, των σχέσεων μεταξύ γειτόνων και να συμπληρώσει τις διμερείς σχέσεις στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, για να ξεπεραστούν οι τοπικές εντάσεις θα πρέπει να εστιαστεί σε πρακτική προσέγγιση και με στόχο με προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Να ολοκληρώσω με λίγες συστάσεις. Επί τη βάση αυτών των συμπερασμάτων έχουμε να κάνουμε τις εξής ε, συστάσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα και αυτό κυρίως σημαίνει ορατή χρηματοδότηση, δηλαδή μια συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού. Δεύτερον, η Ένωση μέσα σε αυτή τη διάσταση, να προσθέσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση την διάσταση της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα με τις χώρες εταίρους. Δηλαδή να ενσωματωθεί αυτή η συνεργασία στις διμερείς σχέσεις ε, να επιστιάσει επίσης περισσότερο σε ένα μικρό αριθμό προτεραιοτήτων ώστε να μην διασκορπίζεται το ενδιαφέρον και φυσικά η η εταιρική σχέση για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό βήμα. Ε, συστηματικά θα πρέπει να προωθεί μια προσέγγιση με βάση προγράμματα. Αυτή ήταν πολύ θετική προσέγγιση και εμπλέκει και την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Να ξεκινήσει εμπλέκοντας ε, περιφερειακούς εταίρους και φορείς ε, στα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού των προγραμμάτων ώστε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον ε, και τέλος ε, θα πρέπει να προσφέρεται μεγαλύτερη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών μας στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα. Οι βασικές συστάσεις λοιπόν αφορούν την παρακολούθηση που βέβαια θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορέσει να, υπάρξει, να υπάρξουν περαιτέρω προσαρμογές πολιτικής και η δεύτερη σύσταση αφορά την ορατότητα. Η συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη ορατότητα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε κυρία Δελκούρ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κάνιχαμ. 10, maximum 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή, κύριε και κύριοι, Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω σήμερα την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Θα ρίξω μια ματιά στο ιστορικό, πρώτα στο ευρύτερο πλαίσιο, μετά στο ιστορικό από τον Αύγουστο 2008. Θα προχωρήσω σε λίγες συστάσεις για βήματα προς τα εμπρός, για την διάρθρωση μιας νέας πολιτικής και θα κάνω και ορισμένα σχόλια καταληκτικά. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε, αλλά ίσως είναι σωστό να το υπενθυμίσουμε, ότι Γνωρίζουμε ότι η ιστορία και η πορεία της περιοχής του Ευξήνου Πόντου μέχρι τώρα είναι διαφορετική. Είναι λιγότερο σημαντικές οι μετασχηματιστικές δυνάμεις από ό,τι στη Δύση. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης άφησαν τις χώρες της περιοχής απροστάτευτες και τρωτές και δημοκρατικά υπανάπτυκτες. Ε, υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να πέσουν υπό την επιρροή ε, κάποιων τοπικών ε, δυνάμεων όπως Τουρκίας και Ρωσίας. Οι δημοκρατικοί θεσμοί εξακολουθούν να αναπτύσσονται στις χώρες αυτές, αλλά έχοντας δυσκολίες να αντιμετωπίσουν εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Πρέπει να προωθηθούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά η κατάσταση όπως είναι τώρα αναγκάζει τους ηγέτες να, της Μαύρης Θάλασσας να παραμένουν μέσα σε κάποιες άκαμπτες ε, σχέσεις αφενός ανάμεσα στη Ρωσία που επεκτείνει την σφαίρα επιρροής της, από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, περισσότερο τώρα διαφυλάσσει τα κεκτημένα παρά ε, προσπαθεί να επεκταθεί. χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των σχέσεων αυτών για χώρες οι οποίες έχουν κίνδυνο και συγκρούσεων. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας έδειξε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πάει πολύ μακριά, χρησιμοποιώντας και βία ενδεχομένως, εφόσον κάποια χώρα προσπαθήσει να ξεφύγει από τη σφαίρα επιρροής της. Υπάρχει και το θέμα της, ε, του ε, ρωσικού στόλου της, ε, του Ευξήνου Πόντου στη Σεβαστούπολη, ανάπτυξη των βάσεών της και χρήση παντό μέσου ε, και οικονομικών δηλαδή. τα, τα, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν κάποιε ε, ανησυχητικές εξέλιξει και αυτέ κάνουν μια ε, περιφερειακή προσέγγιση πιο δύσκολη. Η περιοχή αυτή έχει περάσει από το Αύγουστο του 2008 πολύ σημαντική εξέλιξη αναγκάζοντας έτσι τις χώρες να επαναξιολογήσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ τους, με τις ΗΠΑ, με τη Ρωσία με σημαντικό αποσταθροποιητικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε περιφερειακή στρατηγική προς τον εύξηνο πόντο θα πρέπει να, να την ξανασκεφτεί όποιος θέλει να την ασκήσει. Η οικονομική κρίση έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο επίσης. Έπληξε και την Ευρώπη και την περιοχή τον κόσμο ολόκληρο δηλαδή, εντελώς απρόσμενα και είχε δύο αποτελέσματα για τις χώρες του εύξηνο πόντου. Αφενός αύξηση της ανεργίας, μείωση της εμπιστοσύνης της κυβερνήσης που οδήγησε με τη σειρά της σε, μεγάλες, σε πολλές ε, κοινωνικές αναταραχές. Ο κόσμος χάνει τις δουλειές του, η οικονομία μειώνεται, ε, τα επίπεδα δηλαδή. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να ικανοποιήσουν και τους πολίτες και τους πιστωτές τους. Αναπτύσσεται λοιπόν και άλλο δυναμικό κρίσης. Οι χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης έχουν πληγεί από την κρίση, το ίδιο και ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα και οι κυβερνήσει των Ηνωμένων Πολιτειών και τη ε, Ενωμένη Ευρώπη αντιμετωπίζουν πιέσει από του πολίτε του να στρέψουν τα βλέμματά του περισσότερο προ τα εσωτερικά. Έγινε επαναξιολόγηση και στην Ευρώπη ε, τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ακόμα τώρα αξιολογούνται τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής και ο έξινος πόντο έχει γίνει λοιπόν, λοιπόν λιγότερο, λιγότερο σημαντική προτεραιότητα τώρα. Αφενό οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αφενός μάλλον η Ηνωμένη Ευρώπη. Αφετέρου οι Ηνωμένε Πολιτείε. Με νέα κυβέρνηση που πάτησε το κουμπί reset όπως είπε για τις σχέσεις με τη Ρωσία Δεν έχει καμία συνεκτική πολιτική βέβαια απέναντι στην Ενωμένη Ευρώπη. Έχει και τους αντιπερισπασμούς της ε, η Αμερικανική κυβέρνηση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Η ίδια λοιπόν η περιοχή του Εύξηνου Πόντου είναι μάλλον η πιο στρατιωτικοποιημένη περιοχή κοντά στην Ευρώπη. Αζερβαϊτζάν, αύξηση του στρατιωτικού ε, εξοπλισμού. Ε, Ρωσία, επέκταση στις περιοχές Αφχαζίας και Νότιας Οσετίας και ο αποσταθαπητικός παράγοντας του Νότιου Καυκάσου. Δύσκολη λοιπόν ε, περιοχή και αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προκλήσεις και, στην, ε, και στην έξινο πόντο. Η Ουκρανία και η Γεωργία που ήταν οι πιο σταθερές χώρες έχουν και αυτές αλλάξει δραματικά από την ε, πορτοκαλή επανάσταση όπως λέχθηκε τότε η Γεωργία έχει βιώσει σημαντική δημοκρατική παρακμή η Ουκρανία στρέφεται περισσότερο τώρα προς τον ε, μεγάλο ανατολικό της γείτονα. Ε, τίθεται λοιπόν ερωτηματικό κατά πόσο υιοθετούν ευρωπαϊκές αξίες οι ε, χώρες αυτές. Η Μολδαβία φαίνεται τώρα να έχει περισσότερο μια τέτοια τάση και από τη Μολδαβία μέχρι το Αζερβαϊτζάν υπάρχει βέβαια μεγάλη, μεγάλη απόσταση, είναι τα δύο άκρα. Όπως είπαν οι προλαλήσαντες, η Ρωσία και η Τουρκία παραμένουν σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή και δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε τον ρόλο τους ε, εφόσον μιλούμε για μια στρατηγική. Από τις πιο πολλά υποσχόμενες εξελίξεις είναι η προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας Αρμενίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή ε, κρατείται όμοιρος η Αρμενία στον Αγκόρνο Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε μερικέ συστάσεις για τις μελλοντικέ κινήσεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς αυτό, αλλά ε, χρειάζεται να συμφιλιώσει, αν θέλετε, τις διαφορές ή τις αντιθέσεις μεταξύ των χωρών μελών απέναντι στην περιοχή αυτή. Και αυτό έχει σχέση βέβαια με τι διαφορετικέ σχέσει των χωρών μελών με τη Ρωσία. Πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια συμφιλίωση σε αυτό ε, το θέμα. Η ανατολική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζεται από τι Βρυξέλλε και από όλε τι χώρε μέλη, αν θέλει να, έχει κάποιο, ε, να αποτελέσει κάποιο μετασχηματιστικό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή χρειάζεται να μιλήσει με μια φωνή, κυρίω για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Η ΚΕΠΑ, η οποία είναι ασφαλώ βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, θα δούμε πώ αναπτύσσεται βέβαια σε σχέση με την περιοχή αυτή, εξετάζοντα την οικονομική κρίση, οι ευρωπαϊκέ χώρε πρέπει να προστατευτούν. Πρέπει να αντιμετωπίσουν μάλλον αυτό το φυσιολογικό αντανακλαστικό που έχουν να προστατεύσουν δηλαδή το εσωτερικό του και την ε, ε, εθνική του οικονομία. Που βλέπουμε να οδηγεί σε προστατευτισμό, σε αύξηση τη ξενοφοβία κ.ο.κ. Χρειάζεται λοιπόν να αντισταθούν σε αυτέ τι τάσει οι ε, χώρε μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσέγγιση προς τον έξινο πόντο, και η Black Sea Synergy. Αυτές είναι σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές. Υπάρχει όμως επικάλυψη και σύγχυση. Ακούσαμε ήδη ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Είναι σαφές αυτό αν πραγματικά τα προγράμματα αυτά θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Εάν οι δύο αυτές πρωτοβουλίες ε, παραμείνουν και οι δύο θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση ε, έργου, δηλαδή το τι κάνει η καθεμία. Χρειάζεται πιο ευέλικτες συνεργασίες που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής του εύξηνου πόντου. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, η ενδυμική διαφθορά στις χώρες του εύξηνου πόντου και πρέπει να υπάρξουν ε, ξεκάθαρες επιπτώσεις όταν υπάρχει διαφθορά. Η αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων αυτών στις εθνικές τους κυβερνήσεις ε, πρέπει να, όπως είπα, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, επίσης να ενισχυθεί η ελευθεροτυπία. Είναι ανισχυτική η τάση όλων των χωρών της περιοχής μιας προσπάθειας λογοκρισίας και καταπίεσης των φωνών της κριτικής. Η περιοχή επίσης βέβαια χρειάζεται να αντιληφθεί ότι το μέγα βάρος τον αναλαμβάνουν οι ίδιες να δημιουργήσουν δηλαδή πραγματικά ε, λειτουργικά δημοκρατικά συστήματα. Όπως είπαν οι δύο προλαλήσαντες, είναι πολύ σημαντική η ε, πρόθεση της πολιτιστικής αλληλοκατανόησης στην περιοχή. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να επιληθούν οι φυστάμενες διαφορές, οι παγωμένες συγκρούσεις με την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την βόρεια διάστασή της που έχει κάνει σημαντική κεφαλαιοποίηση από αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες αυτές και για να συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών στον εύξηνο τόπο, στον πόντο. Λοιπόν, σημαντικές, σημαντική μετασχηματίση τα τελευταία χρόνια. Λόγω και του καταλητικού ρόλου της οικονομικής κρίσης παρατείνονται ε, οι περιφερειακές ε, συγκρούσεις ενισχύονται τοπικοί παράγοντες όπως η Ρωσία και η Τουρκία. Οι Ενωμένες Πολιτείες και η Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να διατυπώσουν ξεκάθαρες πολιτικές οι οποίες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της περιοχής. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το μέγα αυτό ιστορικό εγχείρημα της ανατολικής ε, προσέγγισης, της γειτονίας δηλαδή, αν τελικά πηγαίνει να, να φτάσει σε ένα τέλος. Χρειάζεται συγκεκριμένε πρωτοβουλίε υπέρ των χωρών εκείνων που επιθυμούν να υιοθετήσουν ε, δυτικά μοντέλα και δυτικέ αξίε. Η ώρα έχει έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει περισσότερο ηγετικό ρόλο στην ε, περιοχή αυτή γειτονία τη. Έχει τεράστιο δυναμικό η περιοχή του Εύξηνου Πόντου, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Ευχαριστώ κύριε Κάνιχαμ. Αρχίζει η συζήτηση. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να περιορίσω το χρόνο αγόρευσή σας σε ένα τρίλεπτο έκαστος. Ο συνάδελφος Πάσκου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και σκιώδης ηγητής από πλευράς της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Πάσκου. Σίγουρα η περιφέρεια του Ευξήνου Πόντου είναι και σημαντική και σύνθετη, ε, και περίπλοκη. Και ενδεχομένω μπορεί να φορτίσει αρνητικά την ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη. Το έχει κάνει στο παρελθόν και μπορεί και στο μέλλον να συμβεί αυτό. Το ξέρω ότι είναι καλή συνέργεια και συνεργασία. Έχει αποδειχθεί ότι εσφράγισε τη σημασία της περιοχής. Αναγνώρισε δηλαδή ότι η περιφέρεια είναι σημαντική. Αλλά είναι λίγο ιδεαλιστική έτσι γιατί φιλοδοξεί ε, να δημιουργήσει συνοχή ε, γύρω από μια ιδέα που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε. Ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση πριν από 20 χρόνια και ξαφνικά εμείς περιμένουμε να λειτουργεί η περιοχή σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια ή τις δικές μας προσδοκίες για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί μια τέτοια περιφέρεια. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε ταξί τρία προβλήματα. Το πρώτο, τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγική σχέση με τη Ρωσία και οτιδήποτε συμβαίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι σε αυτό το πλαίσιο, σε, σε αυτό και όχι σε τούτο εδώ του ευξήνου πόντου. Και ε, εκεί πέρα δεν ε, υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία ε, συνεργασίας, αλλά μάλλον σύγκρουσης Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες διστάζουν να, μπουν σε ένα παίγνιο πάρα πολύ περίπλοκο και ουσιαστικά συγκρουσιακό στον εύξηνο πόντο. Μετά έχουμε την Τουρκία, άλλο πρόβλημα και τρίτο πρόβλημα η Ουκρανία. Εντάξει. Είναι προβληματική η σχέση τους, αν μη τι άλλο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για στρατηγική, η στρατηγική σημαίνει και προσήλωση, δέσμευση, αφοσίωση. Πόθεν αυτή για να περιμένουμε και στρατηγική. Και κάτι άλλο όμω που είναι ελπιδοφόρο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία να συνεργαστούμε για τη στρατηγική του Δουνάβεως. Και ο Δούναβης χύνεται στον εύξηνο πόντο και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και είναι και στο δικό μας γήπεδο ξέρω και βλέπω εκεί μια θετική ε, διάσταση και ένα δυναμικό που θα μπορούσε να ε, διασπαρεί και προς τον εύξηνο πόντο. Υπάρχει όμως το εξής θεμελιώδες πρόβλημα. Αν για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις σχέσεις τους με την Κίνα, που είναι πάρα πολύ πιθανό για το ορατό μέλλον, πού θα αφήσει αυτό τις σχέσεις μας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και ιδιαίτερα των χωρών που είναι ε, στην παραμεθόριο περιοχή και εκεί είναι η ε, περιοχή του Ευξηνού Πόντου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Πασκού, το, ρόλο, το λόγο έχει ο κύριος Μποστινάρο που είναι εισηγητή για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιφερειακή Πολιτικής. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, από την περιφερειακή προοπτική, εγώ θα αναφερθώ σε κάποια σημεία κλειδιά στην έκθεσή μου. Ε, είναι καταρχήν πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν όλοι οι φορείς, ε, οι παίκτες της περιοχής, Ένωση, κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, γιατί διαφορετικά η στατική αυτή δεν θα είναι ολοκληρωμένη και δεν θα λειτουργήσει. Δύο, είναι θέμα κλειδί επίσης να υπάρχει συντονισμός. Συντονισμός ανάμεσα στις ε, οργανισμούς τους διάφορους θεσμούς ανάμεσα, ε, μέσα στην Ένωση και αυτούς που θα δημιουργηθούν ε, στο μέλλον. Δηλαδή, με ε, οικονομική συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας, κοινοβουλευτική συνέλευση της οικονομικής συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και με τη συνεργασία αυτή. Εγώ να αρχίσω λέγοντας ένα αστιάκι. Μέχρι σήμερα είχαμε συνεργία, συνεργασία Ε, μάλλον συνεργασία για την ενέργεια. Αλλά αντί να έχουμε συνεργασία είχαμε ένα πόλεμο και μια μεγάλη ενεργειακή κρίση. <laughs> Άρα λοιπόν λειτουργεί αυτή η συνεργασία. Μήπως χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε ώστε να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσουμε από μια ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση στην περιοχή. Τρία, συντονισμός ανάμεσα στα προγράμματα υποδομής που υπάρχουν και που αναπτύσσονται μέσα στην Ένωση σε κάθε κράτος μέλος της περιοχής και προγράμματα τα οποία προβλέπονται από τα κράτη-μέλη στις ε, γύρω περιοχές, όπως το πρόγραμμα για τους αυτοκινητόδρομους. Αλλά όχι μόνο τα προγράμματα υποδομής, κυρίως τα ενεργειακά προγράμματα είναι θέμα κλειδί που σχετίζεται με την παροχή ενέργειας προς την Ένωση, αλλά και με την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, διότι τώρα έχουμε επιτάπητος το South Stream, το Ναμπούκο, αλλά φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι να αποκομίσουμε τα διδάγματα από το Nord Stream, από την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Γιατί αν δούμε τα δύο προβλήματα προκύπτει ότι χρειάζεται περιφερειακή συνεργασία και συντονισμός αλλά και συμφωνία σε σχέση με τα βασικά προγράμματα υποδομών και ίσως και ένα περιφερειακό μέσο που να είναι δεσμευτικό ώστε να ε, χειριστεί τα προβλήματα του περιβάλλοντος γιατί η Μαύρη Θάλασσα είναι μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές γύρω από την Ευρώπη, κοντά στην Ευρώπη και μέσα στα ευρωπαϊκά ύδατα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι που να είναι δεσμευτικό ή μόνο ευχολόγια. Γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μόνο διμερείς συνομιλίες, διμερεί μέσα, είτε από μεγάλα κράτη-μέλη της Ένωσης, είτε από πολυμερείς ε, οργανισμούς αλλά στον τομέα τη ενέργεια. Άμα δούμε το αποτέλεσμα όμω είναι προφανέ. Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μια φωνή. Τελική παρατήρηση, Πρόεδρε, όταν μιλάμε για του φορεί. Είμαστε αρκετά προσεκτικοί όταν ορίζουμε το Τουρκία ως λιγότερο προβλέψιμο εταίρο. Να εξηγηθώ πόσο προβλέψιμη είναι η Ευρώπη όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Τικάου, που είναι η συγγήτρια για γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στον τομέα της Επιτροπής, στο, τομέα δραστηριότητα τη Επιτροπής Βιομηχανία. Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η περιφέρεια της ε, Μαύρη Θάλασσα είναι γεωστατηγική σημασία για την ασφάλεια ανεφοδιασμού σε ενέργεια και για τη διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού της, ε, της Ένωσης, γιατί δίνει πρόσβαση στην Κασπία, στην Κεντρική Ασία και μετά από την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ευρω... μέγα ε, παίκτη στι περιοχέ αυτέ. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στη στρατηγική συνεργασία ΕΕ Ρωσίας και τα κοινά του συμφέροντα στην βελτίωση, στην αύξηση μάλλον του, διευ... του εμπορίου και των επενδύσεων. So I would like to draw... Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας λοιπόν στην στρατηγική συνεργασία ΕΕ Ρωσία και τα κοινά του συμφέροντα στην αύξηση του διμερούς εμπορίου και επενδύσεων καθώς και στη διευκόλυνση και απελευθέρωση του εμπορίου μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι έχοντας υπόψη τι νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου και τα νέα, τις νέες ε, το νέο υδροελεκτρικό εργοστάσιο θα ήθελα να υπογραμμίσω τους βασικούς ε, διαφανείς κανόνες για το εμπόριο, τις επενδύσεις καθώς και τις δίκες συνθήκες για την μεταφορά και το εμπόριο της ενέργειας που χρειάζεται να επιβληθούν στην Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή της. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε εκ νέου πως η ασφάλεια της ενέργειας, των εφοδισμού σε ενέργεια βασίζεται στις διαφοροποιημένες πηγές. Και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκου και να ζητήσω κάτι μελη μαζί με τους εταίρους τους να, επιταχύνουν την εφαρμογή του. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας για την ενέργεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για την οποία ο ΠΟΕ αλλά και η συνθήκη για τον ενεργειακό χάρτη προβλέπουν τις βασικές αρχές. Πρέπει να υποστηρίξουμε την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς και τη ρυθμιστική ολοκλήρωση για την Ένωση και όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρας Θάλασσας στην συνθήκη την, ενέργεια, για την ενέργεια καθώς και για την βοήθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Να βελτιωθεί το εμπόριο, μεταφορά του ε, υδρογοναθράκου στην περιοχή, να βελτιωθούν ε, οι, τα τέρμιναλ για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν επιμένω τώρα σε αυτά και στις λεπτομέρειες, αλλά να αναγνωρίσουμε τη σημασία της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και της Επιτροπής για τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τη διοργάνωση της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρη Θάλασσα, και να καλέσουμε την Κομισιό να αναπτύξει μια τέτοια στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα που θα συνοζεύεται από πρόγραμμα δράσης στους τομείς τη συνεργασία για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντα την ε, διασύνδεση και την επικοινωνία, περιβαλλοντική προστασία, ασφάλεια, μετανάστευση και πολιτιστικέ ανταλλαγέ. Σα ευχαριστώ. Καζάκ, εισηγητή, μάλλον συντάξει νομοδότη τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί ομιλητές. Θα περιοριστώ και εγώ στο να παρουσιάσω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θέλω να βάλω και στη γνωμοδότησή μου ξενόμα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι από το 2000 μέχρι το 2008 η περιοχή του Ευξήνου Πόντου ήταν μάρτυρας μιας εντυπωσιακής θεαματικής οικονομικής ανάπτυξης τάξης του 6% ετησίως. Βέβαια, στη συνέχεια με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, το τραπεζικό σύστημα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπέστη μεγάλο στρες και αυτό είχε ολέθρια επίπτωση στις ροές κεφαλαίων προς την περιφέρεια του ευξήνου πόντου. Γι' αυτό θα προτείνουμε οι χώρες που βρέχονται από τον εύξηνο πόντο να φροντίσουν τα οικονομικά τους με πιο αυστηρό τρόπο και με πιο λιτό τρόπο για να μπορέσουν να ε, αναγκάσουν και τις τράπεζές τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι με τη συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει αλλά μπορεί να αποκομίσει και πολύ σημαντικά ωφέλη συνεργαζόμενοι με την ε, ε, οργάνωση για την παρευξήνια συνεργασία. Ε, υπάρχει ένας οργανισμός, και το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, αλλά υπάρχουν ορισμένα θεσμικά όργανα και ορισμένες διατάξεις που πρέπει να βελτιωθούν. Ας πούμε, η Τράπεζα ε, εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξήνου Πόντου, καθώς επίσης και το Συμβούλιο της Παρευξήνιας Συνεργασίας. Ε, στη συνέχεια θα πρέπει επίσης να ομολογήσουμε ότι αυτή η εταιρική σχέση για το περιβάλλον στα πλαίσια της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα είναι πολύ σημαντικό και οι χώρες της περιοχής καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ενέργεια και να εστιάσουν στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και αυτοκινητόδρομοι που να οδηγούν εκεί για να ενταθεί, να αυξηθεί το εμπόριο και οι οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή. Και ένα τελευταίο. Όλα τα κράτη της περιφέρειας σχεδόν είναι μέλη του ΠΟΕ με εξαίρεση δύο και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για να εναρμονίσουμε κάπως το φορολογικό καθεστώς και να ε, σπάσουν και τα φορολογικά και τα τελωνιακά εμπόδια για την ελεύθερη ε, συναλλαγή στην περιφέρεια του ευξηνού πόντου. Και αυτό θα γίνει αν συνεργαστεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις υπάρχουσες ε, δομές τη κυκλοφορική συνέντευξη του ΠΟΕ και του ΠΑΠΣΕΚ. Ευχαριστώ κύριε Κατσάκ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Γιώτοβα, η συγγήτρια της Επιτροπής Αλίας, συντάκτρια γνωμοδότησης. Θα μιλήσει για την αλία στην Εύξηνο Πόντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Είμαι μέλος της Επιτροπής Αλίας Είμαι υπεύθυνη για τον εύξηνο πόντο για τη γνωμοδότηση αυτή που είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια έκθεση. Όπως γνωρίζετε Έξι χώρες βρέχονται ε, από τον εύξηνο πόντο και δύο μόνο είναι μέλη ε, της Ένωσης, Βουλγαρία και Ρουμανία. Είναι πολύ σημαντική η αλληλευτική πολιτική γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε πραγματικά μια στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Όταν μιλάμε για τη λεκάνη αυτή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει ιδιαιτερότητες και προβλήματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστά δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι όλα έχουν παραμείνει σε περιφερειακό επίπεδο. Το καταλαβαίνουν πολύ καλά η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ε, αλλά είναι μέλη της Ένωσης ε, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Γι' αυτό εγώ καλωσορίζω μια πιο μακροχρόνια στρατηγική για την περιφέρεια αυτή. Ιδιαίτερα θεωρώ ότι ο εύξηνος πόντος και η αλία σε αυτή θα πρέπει να βρουν το δρόμο τους και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σήμερα ελάχιστα ε, ε, ή ε, σχεδόν καθόλου δεν ασχολούμαστε με ε, την αλία, με την οικολογία και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό χρειάζεται διεθνή συνεργασία και πιο στενή έτσι ώστε η Ένωση να έχει τους στόχους τους και στην αλία και στη μελλοντική στρατηγική. Θα ήθελα τέλος να προσθέσω την πρόσφατη δημιουργία της κοινοβουλευτικής διάσκεψης ε, η συνέλευση συγγνώμη, της Euronest θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε πλήρως γιατί ε, και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, τίποτα δεν θα είναι εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Αλία, με σημαντικές χώρες γείτονες που είναι η Ρωσία, η Τουρκία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Επιτρέψτε μου να μιλήσω και εξ ονόματος των Αλιαίων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η ίδια τους επιβίωση και το επάγγελμά τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική μας για τον εύξηνο πόντο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόβατζεφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες. Τα συμπεράσματα ήταν ότι χρειάζεται περισσότερη ορατότητα της στρατηγικής του Ευξήνου Πόντου μέσα στα πλαίσια των πολιτικών της Ένωσης και να παίξουμε πιο ενεργό ρόλο. Αυτό θα είναι προ συμφέρον των χωρών μελών τη Ένωση αλλά και προ το συμφέρον των γειτόνων μα. Αυτή η στρατηγική δεν πρέπει να παραμείνει στα χαρτιά. Η Ένωση είναι σημαντική για αυτού, για του γειτονές μας, αλλά και αυτή είναι σημαντική για μας. Η συνεργασία μπορεί να προσφέρει ε, ευημερία και ασφάλεια. Γι' αυτό οι μηχανισμοί της συνέργειας και της ανατολικής γειτονίας πρέπει να λειτουργήσουν εποφελία τους. Και το δημοσιονομικό πακέτο θα πρέπει να δαπανηθεί με τρόπο αποτελεσματικό, γιατί συχνά γνωρίζουμε ότι κυρίως χώρες της κεντρικής Ευρώπης έχουν ε, πρόβλημα απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούω βέβαια πολλά ωραία ρητορικά σχήματα αλλά δυστυχώς πολύ συχνά αποδεικνύονται κούφια λόγια. Ασφαλώς η περιοχή του Εύξηνου Πόντου είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Το γνωρίζω καλά, διότι και η Βουλγαρία βέβαια βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα και μάλιστα και η εκλογική μου περιφέρεια είναι στην Βάρνα. Γνωρίζω πόσο πολύ χρειαζόμαστε την διαμεθοριακή συνεργασία στην περιοχή αυτή. Αυτά που είπε ο κ. Μίντσεφ είναι πολύ σωστά. Και είναι αλήθεια ότι η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει πολλές παγωμένες συγκρούσεις, κυρίως στο ανατολικό μέρος, όχι μόνο τον Κάφκασο αλλά και τον Αγκόνη Καραμπάχ. Εδώ πρέπει να παίξει ενεργότερο ρόλο η Ευρώπη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νέα μας υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας για να διασφαλίσουμε ώστε η Ευρώπη να μην είναι μόνο δωρητής οικονομικής ε, βοήθειας αλλά και να παίξει και ενεργότερο ρόλο σε μια συμβολή επίλυσης των διαφορών αυτών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα είδος brainstorming, δηλαδή να καθίσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς θα βάλουμε μέσα στο παιχνίδι όλους τους φορείς της περιοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόβατσεφ. Ο κύριος Σεβερίν δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες και έχω λίγες ερωτήσεις ελπίζω ε, να μας διαφωτίσουν. Ο τίτλος της ακροάσεως είναι η Ευρωπαϊκή, ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Ε, υπονοώντας ότι δεν αρκεί μια συνεργασία αλλά χρειάζεται μια στρατηγική. Εάν όντως είναι έτσι, μπορούν να μας πούν οι εμπειρογνώμονες ποια είναι η διαφορά μεταξύ της synergy, της συνέργειας δηλαδή και της στρατηγικής. Δεύτερο, Κανονικά μια στρατηγική χρειάζεται μακροπρόθεσμα ζωτικά συμφέροντα. Δεν αναπτύσσει κανεί στρατηγική αν δεν έχει τέτοια μακροπρόθεσμα ζωτικά συμφέροντα. Μπορείτε να μα εξηγήσετε ποια είναι τα μακροπρόθεσμα ζωτικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή. Άλλη ερώτηση. Η Μαύρη Θάλασσα είναι περιοχή ή μάλλον σημείο τομή, σημείο συνάντηση άλλων διαφόρων περιοχών όπου είναι διαφορετικά τα συμφέροντα των διαφόρων δυνάμεων στις περιοχές αυτές. Και τελευταίο, Ρωσία και Τουρκία είναι ξεκάθαρο και από τη δική μου προσωπική εμπειρία κάθε, που, κάθε φορά που προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τους διαφόρους φορείς βλέπουμε Ρωσία και Τουρκία να είναι πολύ διστακτικές να προσέλθουν σε τέτοιες συναντήσεις. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κινητοποιήσει τις χώρες αυτές να αλλάξουν θέση. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν. Ο κύριος Αγκουράκης. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δυστυχώς μέχρι τώρα η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ ευρωβουλευτών που προέρχονται από τον χώρο του Εύξηνου Πόντου, είναι κοντά σε αυτόν. Ελπίζω στη συνέχεια να υπάρχουν και από άλλες περιοχές, γιατί όντως η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πριν να σημειώσω δύο-τρία ζητήματα, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, με όλο το σεβασμό και ε, την εκτίμηση που σας έχω. Έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς οι, οι δύο εισηγητές σήμερα, ειδικοί ο κύριος Μίντσεφ και ε, ο κύριος, ο κύριος Κάνιγκαμ, ελάχιστα μας βοηθήσαν στο να κατανοήσουμε καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα έλεγα, ειδικά ο κύριος Κάνιγκαν διατρέχεται από προκαταλήψεις όσον αφορά τους λαούς της περιοχής και τις χώρες αυτές και επίσης υπάρχουν αρκετές προκαταλήψεις και ανακρίβειες και στην τοποθέτηση του κυρίου ε, Μίντσεφ. Κατά την άποψή μου ήταν μια έκθεση ιδεών για γεωστρατηγικές εξελίξεις οι οποίες είναι τέτοιες ή αλλιώτικες. Ε, θα περίμενα να υπήρχε μια μεγαλύτερη αναφορά ε, σε μια εμπειρία που υπάρχει ήδη από την παραφυξήνια ε, συνεργασία και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους που τοποθετηθήκαν στα ζητήματα αυτά και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Ντελκούρ η οποία ε, μας φώτισε και μας ε, έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις. Δύο ζητήματα μόνο και τελειώνω. Ε, δεν είναι αλήθεια ότι η συνθήκη του Μοντρέ, πώς το λένε, δημιουργεί προβλήματα σαν για αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Μίντσεφ και δεν κατάλαβα πολύ καλά τι εννοεί. Εννοεί δηλαδή να αλλάξει η συνθήκη του Μοντρέ και να αντικατασταθεί από τι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά την, τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ε, μίλησε για μονοπόληση. Γιατί μονοπόληση κύριε Μίντσεβ. Ελεύθερη αγορά υπάρχει, α πάνε οι χώρε να αγοράσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από όπου θέλουν. Είναι άλλο θέμα τώρα ότι η γειτονίαση με τη Ρωσία κάνει τα πράγματα αυτά πιο οικονομικά. Ε, τι να κάνουμε. Να πάμε αλλού, να αλλάξουμε γεωγραφική θέση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Ο εισηγητής ζήτησε να παρέμβει για να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στους εμπειρογνωμονές μα. Δύο λεπτά, γιατί έχετε και το χρόνο στο τέλο. Ναι, θα είμαι σύντομο Πρόεδρε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Νομίζω πως θα πρέπει να έχουν ε, την ευκαιρία οι εμπειρογνώμονές μας να μιλήσουν, στο τε... να απαντήσουν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όντως ακούσαμε πολλά και διάφορα για τη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, είναι μαύρη στα αλήθεια. Είναι μια ρεαλιστική εικόνα αυτή η άποψη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω από τους ε, συζητητές είναι το εξής. Η Μαύρη Θάλασσα μετατρέπεται σε νεκρή θάλασσα ή ξεχασμένη θάλασσα. Δηλαδή η, Μαύρη Θάλασσα είναι περισσότερο ρωσική και τουρκική, δηλαδή τη χάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πριν καν την κερδίσουμε. Δεύτερον, γιατί ακούσαμε τους πυρογνώμονες και τους συναδέλφους να λένε όλο για το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Είναι μία πρόταση, ερώτηση για την Κομισιόν. Τι γίνεται με την ξεκάθαρη χρηματοδότηση για τη Μαύρη Θάλασσα. Και να προσθέσω μία μόνο λεπτομέρεια. έχω δίκιο. Φέτος ε, την Άνοιξη λήφθη απόφαση της Κομισιόν που ανακατένει με 1,5 δις από ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το περιβάλλον στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Σε ένα άλλο πρόγραμμα είστε για τα μπανάνα στις χώρες ΑΚΕ. Τα μετέφερε από τη Μαύρη Θάλασσα στην Πανάνα. Mm. Αυτά θέλω να ακούσω τις απαντήσεις των ε, εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Πριν να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες θα ήθελα να δώσω χώρο, πάλι βέβαια περιορισμένο, στον δόκτωρ Μπεσέ που αντιπροσωπεύει την Κομισιόν για τρία λεπτά για τα δικά του σχόλια. Όπως γνωρίζουμε η ε, Κομισιόν θα έχει τον τρόπο να εμβαθύνει όταν θα συζητηθεί η έκθεση. Άρα λοιπόν το χρόνο που σας ε, κόβω τώρα θα σας το δώσω ε, με το παραπάνω στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως ε, τρία λεπτά για να σχολιάσουμε τα όσα υπόθηκαν είναι μάλλον πνευματικό μαρτύριο παρά οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε κάποια βασικά σημεία. Το πρώτο, και πιστέψτε με, δεν θέλω να είμαι ευγενικό μαζί σας. Το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συζήτηση συμπεριτοχική σήμερα, αυτή την ακρόαση, είναι εξαίρετο νέο. Γιατί για μας πριν από λίγο χαρτολογούσαμε τον εισογητή πριν από την ε, έναρξη τη ακρόαση και του λέγαμε ότι εκείνο δεν με χρειαζόταν, αλλά ότι εγώ τον χρειαζόμουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αν το Κοινοβούλιο δείξει ενδιαφέρον και δυναμισμό ε, στην προσέγγιση του θέματος της Μαύρης Θάλασσας μπορούμε να κάνουμε τεράστια πρόοδο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι για να επανέλθω λίγο στα όσα είπε η κυρία Ντελκούρ σε σχέση με την εφαρμογή της συνεργασίας για τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι μια εφαρμογή που χρονοτριβεί, είναι χαοτική και οι λόγοι που δώσατε οι εξηγήσει που δώσατε εσεί, κυρία μου, είναι σωστέ. Υπάρχουν εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντε. Δεν χρειάζεται τώρα να επεκταθούμε σε αυτό. Αλλά είναι σαφέ και εδώ ήδη φτάνω στην τρίτη μου παρατήρηση. Ό,τι και αν κάνουμε για το θέμα αυτό, εάν προσανατολιζόμαστε προς την επεξεργασία μιας στρατηγικής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ε, φτιάξουμε ακόμα μια φορά ένα υπέροχο έγγραφο το οποίο όμως θα μείνει νεκρό γράμμα και το Κοινοβούλιο ως Δημοσιονομική Αρχή έχει πολύ κρίσιμο ρόλο να παίξει. Μην σταματήσετε στην εκπόνηση ενός εγγράφου. Εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ ότι δεν θα σταματήσουμε στην εκπόνηση του, του, του έγγραφου. Μόνο που έχουμε ανάγκη από μέσα, όχι μόνο χρήματα, χρειαζόμαστε και ανθρώπους, αλλά και ε, πολιτική συγκέντρωση και ενέργεια που να προέρχεται απ' έξω και από μέσα από την Ένωση για να φτιάξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να το υλοποιήσουμε. Ανάμεσα στους παράγοντες ε, που δημιούργησαν το χάος που αναφέραμε πριν είναι προφανές ότι ο πολλαπλασιασμός προγραμμάτων ε, και πρωτοβουλειών που κάθε φορά ζητούν βεβαίως συγκέντρωση όχι μόνο χρημάτων όπως είπα αλλά κονδυλίων δεν βοηθά αυτό στην συνέχιση και στη συνέπεια σε τέτοιου είδους ε, προσπάθειες. Για να μείνουμε στο θέμα τώρα της στρατηγικής. Άκουσα τον εισηγητή, πιστεύω και άκουσαν και τα μέλη που υπογράμμισαν την περιπλοκότητα της περιοχής. Πιστεύω πως κάθε φορά που λέμε δημόσια ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούμε προβλήματα για τους εαυτούς μας. Ε, δεν λέω πως η Μεσόγειο δεν έχει, δεν έχει προβλήματα, αλλά η ιστορική παρουσία της Ευρώπης στη Μεσόγειο είναι διαφορετική. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει από τις Βρυξέλλες μέσα στη Μαύρη Θάλασσα και βουτάει, δημιουργεί ένα πρόβλημα, πρόβλημα ε, ψυχολογικό που δεν θα το έλεγα ότι είναι τείχος, δεν ορθώνεται κάποιο τείχος, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Υπόψη στο λόγο μας, στην επιλογή των μέσων που προτείνουμε. Όλα αυτά λοιπόν για να πω με λίγα λόγια πρόεδρε γιατί βλέπω ότι ο χρόνος έχει δηλήξει. Για μα είναι λοιπόν εξαίρετο το νέο να γίνεται λόγος για στρατηγική, να λειτουργήσουμε με ε, συνεπή και συνεκτικό τρόπο από πολιτική άποψη, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή, τα θα δημιουργήσουμε όλα τα εργαλεία που θα μα χρησιμεύσουν. Είμαστε στη διάθεσή σας για τον εισηγητή και για ολόκληρη την Επιτροπή για να το συζητήσουμε περισσότερο όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπεσέ. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στους εμπειρογνώμονές μας. Είναι δύσκολο να μπορέσουν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις που άκουσαν, αλλά σας παρακαλώ, δεδομένων των ικανοτήτων σας, να το πράξετε αυτό στα 10 λεπτά που μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της ε, συνάντησης. Η σειρά παρέμβασης θα είναι η, ίδια όπως στην αρχή. Θα δώσω το λόγο σε εσά, ε, κύριε Μίντσεφ, πρώτα. Μοιραστείτε το χρόνο σας, 3-4 λεπτά έκαστος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος εγώ όσο μπορώ. Η διαφορά ανάμεσα στη συνέργεια και τη στρατηγική, ή τη συνεργασία και τη στρατηγική η συνέργεια για τον εύξηνο πόντο ήταν μια εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια. Γι' αυτό βασίστηκε σε ένα θεσμικό ε, πλαίσιο που υπήρχε ήδη στον ΠΙΣΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεχωριστός παράγων ε, με, μεγάλη, με επιρροή, με ίδια συμφέροντα που έρχεται ε, στην περιοχή και είναι και σε ανταγωνισμό αν θέλετε ε, με τις άλλες δυνάμεις της περιοχής για να έχει και επιρροή μακροπρόθεσμη. Ποιο είναι λοιπόν το ζωτικό συμφέρον και το μακροπρόθεσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μια τέτοια στρατηγική προς τον εύξηνο πόντο. Είναι μόνο το γεγονός ότι είναι μέλη της ε, η Ρουμανία και η Βουλγαρία και βρέχονται από τον εύξηνο πόντο. Όχι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πάρα πολύ μακροπρόθεσμα και πρόπτικα να έχει μια γειτονία προς Ανατολάς που σε όρους κοινωνικούς και πολιτικούς να αναπαράγει τις περισσότερες αξίες και θεσμικές πρακτικές της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε η γειτονία να είναι φιλική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς θα έχουμε γείτονε που θα καταναλώνουν χρήματα, προσπάθειες και θα χρειάζονται και θυσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πρόκειται για χώρε που μπορεί να γίνουν κάποτε μέλη τη Ένωση ή και ποτέ, το μακροπρόθεσμο συμφέρον είναι να δημιουργήσει ένα εξωτερικό κύκλο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να είναι ας πούμε μια κοινοπολιτεία κρατών με ευρωπαϊκούς όρους και να ανήκει στις αξίες και στις αρχές της Ένωσης και στο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να είναι για κάποιο χρονικό διάστημα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε. Και η περιοχή του Ευξήνου Πόντου, κατά την άποψή μου, μπορεί να θεωρηθεί μια ολόκληρη περιφέρεια που με κάποιο τρόπο ανήκει στην Ευρώπη και στα βροδρόμια διαφόρων πολιτισμών και διαφόρων στρατηγικών παραγόντων. Όπως και να θεωρούμε πάντως την περιφέρεια αυτή, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παράγοντας πρωτογενού σημασίας, πρωταγωνιστής στην περιοχή. Οι άλλες δυνάμεις και του status quo, η Ρωσία και η Τουρκία θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, αλλά μην τους εκχωρήσουμε και την ηγεμονία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταλκούρ. Τρία-τέσσερα λεπτά παρακαλώ κι εσείς. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κυρίως τώρα για τρία σημεία εγώ. Το θέμα της στρατηγικής για μένα η στρατηγική θα είχε δύο βασικές ε, λειτουργίες. Να αυξηθεί η προβολή, η ορατότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια και με δραστηριότητες και πρωτοβουλίες όπως είναι η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Γειτονία. Να μην γίνει μια ξεχασμένη περιφέρεια η Μαύρη Θάλασσα. Το δεύτερο ενδιαφέρον αυτής της στρατηγικής θα ήταν ότι θα προσδιορίζε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια που βεβαίως είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα που να βασίζεται ακριβώς στο ότι συμμεριζόμαστε κάποιες κοινέ αξίες. Σε ό,τι αφορά τη συνέργεια, τη συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκε το σχόλιο ως προς τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία των περιοχών Μα ακριβώς εκεί έγκυται και η υπεραξία ή το κέρδος. Συνδέονται διάφορες περιφέρειες και ανοίγουμε καινούργιες πόρτες προς την Κεντρική Ασία και την Κασπία. Είναι ένα μοναδικό ε, μέσο και εργαλείο αυτό γιατί ε, συνεργάζονται έτσι χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Για τη Ρωσία, πώς να την ενθαρρύνουμε. Ε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ερώτηση. Μα αυτό βρίσκεται στην ίδια τη ρίζα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χώρες που είχαν στο παρελθόν τεταμένες σχέσεις, στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν, πώς θα μπορέσουν να συνεργάζονται. Ε, αυτό τίθεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς μπορούν να συνεργαστούν διάφορες χώρες με τη μέθοδο των μικρών βημάτων του Ζαμονέ και με συγκεκριμένη συνεργασία. Εξού και η εταιρική σχέση και η συνεργασία για το περιβάλλον, ας πούμε, που μόλις ξεκίνησε. Είναι πολύ συγκεκριμένες μέθοδοι που έχουν αποδείξει ε, ε, τη σημασία τους και την αποτελεσματικότητά τους σε άλλο επίπεδο, στη βόρεια ευρωπαϊκή διάσταση, συνεργασία με τη Ρωσία βέβαια είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά αποδίδει. Η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο βασικοί συνομιλητές ε, στη Βαλτική, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν πολύ περισσότεροι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντελκούρ. Τα τελευταία τρία λεπτά είναι για τον δόκτορα Κάνιχαμ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διόλου δεν ήθελα να περάσει ένα απεσιόδοξο μήνυμα. Προσπαθούσα περισσότερο να δώσω ένα νέο πλαίσιο για την άσκηση πολιτικής. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Μπεσέ ότι είναι ε, πολύ σημαντική η συζήτηση που γίνεται σήμερα και καλοδεχούμενη για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για την περιοχή πρέπει να πάρουμε υπόψη το ε, οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα. Εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι η συνέργεια για τον εύξηνο πόντο ήταν καλή αφετηρία. Έγιναν πρόοδοι στην περιοχή αυτή, προώθηση συνεργασίας σε διαφόρους τομείς όπως το περιβάλλον, η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, η ε, χρήση των υδάτων, ορισμένες συνεργασίες στην ναυτιλιακή ασφάλεια, επιμέρους δηλαδή περιφερειακής συνεργασίας, χωρίς να ανατραπούν οι συσχετισμοί δυνάμεων. Δεν πάει να γίνει ο εύξηνος πόντος λησμονημένη θάλασσα, ούτε πρόκειται να τη χάσουμε πριν να την κερδίσουμε. Ε, οι δύο μηχανισμοί που υπάρχουν ήδη αποτελούν σωστή αφετηρία. Αλλά πρέπει να λάβουν υπόψη το νέο πολιτικό πλαίσιο και πρέπει να δομηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αρκετά εύκαμπτοί για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ε, διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιοχής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κάνιχαμ. Τελικά συμπεράσματα και σχόλια από πλευράς του εισηγητού κ. Ουγγουρεάνου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ και για τα σχόλια των συναδέλφων. Τι να προσθέσω άραγε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και άλλη ακρόαση. Άλλη διαφορετική. Πάντως νομίζω ότι έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που βρίσκεται η κατάσταση στην ε, περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και πράγματι μπορούμε να συμπεράνουμε όντως ότι η Μαύρη Θάλασσα δεν πρόκειται να γίνει μια λησμονημένη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι εάν η Μαύρη Θάλασσα δεν, πρέπει να, δεν κινδυνεύει να λησμονηθεί Άραγε ε, λόγω των όσων, κάνουν, των όσων κάνουν άλλοι παράγοντες εκεί και όχι των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαύρη Θάλασσα είναι περιοχή κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι περιφερειακή από στρατηγική και ενεργειακή άποψη. Λοιπόν, από στρατηγική και ενεργειακή άποψη είναι κεντρική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα που ακούστηκε καθαρά σήμερα είναι η ανάγκη ανάπτυξης μιας ιδιαίτερης στρατηγικής όπως είπαν και οι πάνελιστ υπάρχει πραγματικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο μείζον θέμα που τέθηκε σήμερα ήταν το χρηματοδοτικό που αποτελεί μέρος του γενικότερου προβλήματος που αναφέρεται στην ανάγκη να δημιουργηθούν ρεαλιστικοί μηχανισμοί και πολιτικές για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιοχής του εύξηνου πόντου. Ξέρω ότι κάπως έχουμε καθυστερήσει. Εκφράζω λοιπόν και πάλι <clears throat> τις ευχαριστίες μου σε όλες και όλους όσοι συμμετέσχουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συζήτηση το συντομότερο δυνατόν. Σα ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Όλους όσου συμμετείχατε, τους εμπειρογνώμονέ μας, τον Δόκτωρ Πεσέ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα εμβαθυνθεί όταν ε, θα είναι έτοιμη η έκθεσή σα, κύριε Γκουεράνου. Η επόμενη μας ε, ε, συνεδρίαση είναι στις 20 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Ναι.